Ο πρόεδρος. Καλημέρα σας. Παρακαλώ καθίστε, αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακαλώ καθίστε. Άρχεται η συνεδρίαση, οπότε σας παρακαλώ καθίστε. Άρχεται λοιπόν η συνεδρίαση. Καταρχά έχω αίτημα του κυρίου Γκόλνη για διαδικαστικό θέμα. Παρακαλώ κύριε Γκόλνη. Το μικρόφωνο μου λειτουργεί. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Το διαδικαστικό μου βασίζεται στο άρθρο 118 του κανονισμού που αφορά την ακρόαση που έγινε χθες για τους υποψηφίους επιτρόπους στην Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών και Εξωτερικών Υποθέσεων έγιναν διακρίσεις που νομίζω ότι είναι αντίθετες προς τον κανονισμό. Δηλαδή δεν δόθηκε λόγος στους μη εγγεγραμμένους. Το άρθρο 118 που ρυθμίζει το θέμα αυτό παραπέμπει στο, παρά, στο παράρτημα 16 το οποίο προβλέπει ότι αν οι συντονιστές των ομάδων έχουν μεν αρμοδιότητα για την οργάνωση της συζήτησης αλλά ο χρόνος ομιλίας κατανέμεται ανάλογα με το άρθρο 162 το οποίο στην παράγραφο 4 προβλέπει και επανειλημμένα χρόνο ομιλίας για τους μη εγγεγραμμένους. Άρα υπήρξαν διακρίσεις και ελπίζω να μην προαγγέλουν τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ελέγξουμε και θα σας ενημερώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν περάσουμε στην ημερήσια διάταξη, Καταρχάς, σύντομα θα ήθελα να ε, πιστήσω την προσοχή σας σε ένα συνάδελφο που κάθεται εδώ αριστερά μου ο οποίος για πολλές δεκαετίες φρόντισε για να λειτουργήσει με ορθό τρόπο το Κοινοβούλιο και Ολομέλεια. Ο κύριος Πολ Ντάνσταν είναι τελευταία ημέρα που εργάζεται για μας κύριε Ντάνσταν υπηρετήσατε το σώμα μας για δεκαετίες ήταν υπεύθυνος για διεξαγωγή εξαγωγή της ολομέλειας του σώματός μας